πια. <clears throat> Κυρίες και κύριοι, ξεκινάμε. Προεδρεύω μετά από αίτημα της απερχομένης Προέδρου ως παλαιός αντιπρόεδρος. Είναι διαθέσιμες όλες οι γλώσσες στη διευμηνία εκτός από τα μαλτέζικα, που έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι δεν έχουμε βουλευτεί από τη Μάλτα. Θα ήθελα να καλωσορίσω λοιπόν όλα τα μέλη της Επιτροπής Τραν. Ε, θα συνεργαστούμε τα επόμενα χρόνια. Θέλω επίσης να καλωσορίσω και τα παλαιά μέλη, τα οποία με χαρά συναντώ εκ νέου. Στόχος της συνεδριάσεώς μας είναι η εκλογή της, του Προέδρου και των τεσσάρων αντιπροέδρων. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με την εκλογή της του Προέδρου και μετά θα με διαδεχθεί εδώ για να συνεχίσουμε τις υπόλοιπες εκλογές. Υπάρχει απαρτία, όμως σύμφωνα με τον κανονισμό οφείλω να σας ενημερώσω ότι κάποια πλήρη μέλη ε, δεν μπορούσαν να είναι εδώ και αντικαθίστανται με συμφωνία της ομάδας τους από αναπληρωτές. Θα σας διαβάσω τον κατάλογο εφόσον δεν υπάρχει κάποια αντίρρηση. membre titulaire PPE est remplacé par M. Tomasz Frankowski. Madame Karima Deli, seulement pour l'élection à la présidence, sera remplacée. Μόνο για την ε, εκλογή για την Προεδρία η κυρία Ντελή θα αντικατασταθεί από την κυρία Ντάουλινγκ. Η κυρία Τίλιβερ για τους πράσινους θα αντικατασταθεί από τον Ντάνιελ Φρόιντ. Ο κύριος Κάμπο Μετσόνη για την ID θα αντικατασταθεί από την κυρία Χάιντερ. Ο κύριος Προέμπα θα αντικατασταθεί από τον Άντζελ Τσαμπάσκι. Ο κύριος Ζωάου Φερέιρα για την ΚΟΕ αντικαθίσταται από την κυρία Αν Πελτιέ η κυρία Κατερίνα Κονέτσνα αντικαθίσταται για την ΚΟΕ από την κυρία Κλέα Ντάλι και ο κύριος Ντέιβιν Μπάουλ των μη εγγεγραμμένων αντικαθίσταται από τον κύριο Ουέλς. Αν δεν υπάρχει κάποια παρατήρηση θα ξεκινήσουμε αμέσως τη διαδικασία ψηφοφορίας. Παρακαλώ έχετε όλοι βεβαιωθείτε την κάρτα σας, αν και δεν θα είναι υποχρεωτικά ηλεκτρονική η ψηφοφορία, αλλά Καλό θα είναι να την έχετε έτοιμη, έτσι ώστε να μην χάσουμε χρόνο. Καλώς. Θα ήθελα λοιπόν τώρα να ζητήσω ε, τα ονόματα ε, για την Προεδρία της Επιτροπής Μεταφορών. Ποιος είναι υποψήφιος για την ομάδα των Πρασίνων θα ήθελα να προτείνω την κυρία Ντελή. Ευχαριστώ πολύ λέει ο πρόεδρος. Υπάρχουν άλλες προτάσεις, άλλες υποψηφιότητες. Όχι. Ζητώ από την κυρία Ντελή να μου πει αν δέχεται την υποψηφιότητα. Κύριε Ερικέ, δέχομαι με χαρά την υποψηφιότητά μου. Σύμφωνα τώρα με τα κοινοβουλευτικά ήθη, εφόσον δεν υπάρχουν άλλοι υποψήφοι, θα ήθελα να εκλέξουμε διαβοή στην κυρία Ντελή. Madame la Présidente, je vous invite à siéger et je vous cède la place. chers collègues. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε και κύριοι, ευχαριστώ τον Ντομινίκ Ρικέ, δεν είναι ένα βουλευτή σαν όλου, του άλλου. ήταν ο πρώτο αντιπροεδρό μου τα τελευταία δυόμιση χρόνια, είναι ένα φίλο, είναι ένα γνώμων. είναι βασικό τέλεχος τη Επιτροπή Μεταφορών. Να ευχαριστήσω όλου του παλαιού συναδέλφου τα τελευταία χρόνια, να καλωσορίσω τα νέα μέλη, άνδρες και γυναίκες, αυτής εδώ της Επιτροπής. Είμαι ιδιαίτερα υπερήφανη για την επιλογή μας. Είναι σημαντικό που εκλέξατε μια νέα γυναίκα στη θέση αυτή, στέλνετε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους Ευρωπαίους πολίτες. Εγώ ποτέ δεν πίστευα ότι θα ξαναείμαι εδώ πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών, που για μένα έχει μεγάλη σημασία. Είναι μεγάλη τιμή για μένα, αλλά ταυτόχρονα είναι και κάποια ευθύνη να αντιμετωπίσω την πρόκληση μπροστά μας, αλλά την πρόκληση ακριβώς της νεολαίας την οποία υποδεχθήκαμε εδώ και λίγους μήνες που είχε ζητήσει ένα πράγμα να πάρουμε τις ευθύνες μας, να αναλάβουμε τις ευθύνες μας έτσι ώστε το κατεπήγον θέμα του κλίματος και του περιβάλλοντος να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Ο τομέας των μεταφορών έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Έχουμε την μεγάλη ασθένεια του 21ου αιώνα, τη μόλυνση που σκοτώνει χιλιάδες ανθρώπους κάθε χρόνο και τα μέτρα δεν λαμβάνονται υπόψη, δυστυχώς δεν λαμβάνονται καν ε, σε σωστό χρόνο με πολλές συνέπειες. Τώρα ε, η αποστολή μας είναι ξεκάθαρη να διευκολύνουμε τις μεταφορές, να διευκολύνουμε την κινητικότητα, να διευκολύνουμε τις μετακινήσεις για όλους, να σεβαστούμε το περιβάλλον και να δώσουμε σε όλους εγγυήσει για μια θέση απασχόλησης υψηλής ποιότητας. Αυτή είναι η αποστολή μας υψηλού επίπεδου εγώ θα είμαι πάντα στη διάθεσή σας, η πόρτα του γραφεία μου θα είναι πάντα ανοιχτή. Βλέπω εδώ και τη γραμματεία, ξέρω ότι δεν είναι απλοί γραφειοκράτες, είναι εμπειρογνώμονες. Υπηρετούν τους βουλευτές οι άνθρωποι αυτοί. Και εσείς λοιπόν έχετε πολύ σημαντικό ρόλο ε, η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση έχει ανάγκη τη συμμετοχή όλων, το πακέτο κινητικότητας. Δώσαμε μάχες ε, για να το διαπραγματευτούμε. Κύριε Μαρινέσκου πρέπει να το ολοκληρώσουμε πλέον. Και ε, μπορείτε να υπολογίζετε σε μένα, θα έχουμε ένα πρόγραμμα φιλόδοξο, θα συζητήσουμε με το Συμβούλιο και την Επιτροπή στα πλαίσια των τριμερών διαλόγων και ελπίζω να πετύχουμε την ίδια σωστή δυναμική με την προηγούμενη εντολή. Και θα πρέπει επίσης να ακολουθήσουμε και αυτά τα οποία είχε πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου και στον τομέα των θαλασσίων μεταφορών της ναυσιπλοείας θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε ε, στα υπεροκεάνια, στα κρουαζιερόπλια, νέες συνθήκες ασφαλείας γιατί και ο τουρισμός ανήκει στις αρμοδιότητές μας. Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα έτσι ώστε η ψηφιοποίηση και η καινοτομία να χρησιμοποιηθούν στον μέγιστο βαθμό. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε δυναμική και σε κοινωνικούς κανόνες που να απαγορεύουν το κοινωνικό dumping, έτσι ώστε η Ευρώπη να λειτουργήσει κοινωνικά και τελειώνοντας με μια σημαντική παρατήρηση νομίζω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πύλη μέσα από την οποία ο πολίτης θα έρθει στην Ευρώπη. Γι' αυτό ακριβώς ε, θα καλούμε στα πλαίσια των λεγόμενων ε, συναντήσεων με τους πολίτες ε, της αγοράς επικοινωνίας θα έλεγα και στον τομέα της κινητικότητας τηρώντας την δεοντολογία. Εγώ πρόεδρος αναλαμβάνω την ευθύνη όπως και όλοι σας να υπογράψουμε την χάρτα επίσης και για τα οικονομικά συμφέροντα. Η αναγνωσιμότητα και η διαφάνεια θα πρέπει να μας χαρακτηρίζει. Τελειώνοντας ότι αυτή εδώ επιτροπή και είναι σαφές και στρέφομαι στον κύριο Μαρινέσκου ε, θα διαπραγματευτεί ε, σκληρά με το Συμβούλιο και την Επιτροπή έτσι ώστε οι θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να μεταφέρονται πάντα σωστά. Η Επιτροπή είναι θα έλεγα υποχρεωτικός εταίρος στις συζητήσεις αυτές και θα είμαστε βασικός πυλώνας σε τομείς ε, στους οποίους πολλές προσπάθειες πρέπει να γίνουν και να επανέλθουμε σε συγκεκριμένες προτάσεις. Ελπίζω να πετύχει η αποστολή μας. Θα ξεκινήσουμε αμέσως με την πρόταση ε, για τη σύσταση του Προεδρείου της Επιτροπής. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν να ζητήσω αν υπάρχει υποψήφιος για τον πρώτο αντιπρόεδρο στο εσωτερικό της Επιτροπής μας, ο κύριος Λιμπεράτσκι. Έχετε το λόγο. Thank you very much, dear Karima. Ευχαριστώ αγαπητή Καριμά και συγχαρητήρια για την εκλογή σου διαβοής. Καλές ειδήσει είναι αυτές, αλλά έχουμε και συνέχεια. Μίλησες πάρα πολύ ε, για την αποστολή μας για τις μεταφορές, δεν είναι μόνο αρνητικά στις μεταφορές, θέλω λίγο να βάλω μια απόχρωση εδώ. Ε, είναι και θέσεις εργασίας, είναι και επιχείρηση, ε, ε, οι μεταφορές και ποιότητα ζωής και οικονομική ανάπτυξη. Προτείνουμε ως πρώτο αντιπρόεδρο το συνάδελφο των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, το Σουηδό Γιώχαν Ντάνιελσον, που προέρχεται από τα συνδικάτα γιατί είναι πολύ σημαντικές οι δουλειές και οι ποιοτικέ δουλειές. Εκατομμύρια ε, ανθρώπων απασχολούνται στις μεταφορές και βγάζουν το ψωμί τους από εκεί. Και προτείνουμε και τρίτο αντιπρόεδρο σοσιαλιστές και δημοκράτες, τον Ιστφαν Ιχελή, ο οποίος έχει πολύ μεγάλη πείρα στις επιχειρήσεις εκεί, για να έχουμε και μια πολύ καλή γεωγραφική ισορροπία. Δύο ονόματα προτείνουμε λοιπόν, σοσιαλιστές και δημοκράτες, για τον πρώτο και τον τρίτο αντιπρόεδρο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Άλλος υποψήφιος. Κύριε Ντάνιελσον, δέχεστε την υποψηφιότητά σα. αυτή. Dear colleagues, I'm delighted to accept Με πολύ μεγάλη χαρά, ευχαριστώ. Είμαι πανευτυχής. Ευχαριστώ κύριε Ντάνιελσον. Εάν δεν έχουμε άλλο υποψήφιο για τη θέση του πρώτου αντιπροέδρου, ψηφίζουμε. Δια Ελάτε κύριε Ντάνιελσον στο Προεδρείο σας παρακαλώ, ως πρώτος αντιπρόεδρος πλέον. Et nous Και συνεχίζουμε. Δεύτερος αντιπρόεδρος. Έχουμε υποψηφιότητα. Ο κύριος Μαρινέσκου ζητεί το λόγο. Παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, σας προτείνω από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα τον κύριο Σβέν Σούλτσε. Άλλον υποψήφιο έχουμε. Όχι. Κύριε Σούλτσε, δέχεστε. Αποδέχεστε την υποψηφιότητα. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την πολιτική μου ομάδα για την υποψηφιότητα. Σήμερα δεν υπάρχει τίποτα ωραιότερο από το να είναι κανείς υποψήφιος για να μπορεί να έρθει να παρακαθίσει εκεί στο Προεδρείο κοντά σας. Οπότε με πολύ χαρά δέχομαι αυτή την ε, πρόταση. Προτείνω λοιπόν διαβόηση επίσης. Συγχαρητήρια κύριε Σούλτσε. Θα είστε το νούμερο δύο μου. Ελάτε. Continuons. Συνεχίζουμε τρίτος αντιπρόεδρος. Κύριε Λιμπεράτσκι. Ναι, σας είπα προηγουμένως ότι πρότεινα τον Ιστβαν Βίχελη για τρίτο αντιπρόεδρο. Με μεγάλη μου χαρά επαναλαμβάνω την υποψηφιότητα και σας ζητώ να τον υποστηρίξετε και να τον εκλέξουμε διαβοής. Αν δεν έχουμε άλλο υποψήφιο, θα ρωτήσω τον κύριο Ουίχελη Συμφωνείτε με την ε, πρόταση αυτή για να γίνετε ο τρίτος μου αντιπρόεδρος. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Thank you so much, colleagues. It is my big pleasure. Σας ευχαριστώ. Με πολύ μεγάλη μου χαρά για να υπηρετήσω τον τουρισμό και τις μεταφορές και την οικογένεια αυτή εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Εφόσον δεν υπάρχει άλλος υποψήφιος, διαβοή και αυτή η εκλογή, παρακαλώ, ελάτε και εσείς εδώ στο Προεδρείο κοντά μου. Για τον τέταρτο αντιπρόεδρο τώρα έχουμε υποψηφιότητες. Thank you on ID Εξ ονόματος της ομάδας ID, Ταυτότητα και Δημοκρατία, θα ήθελα να προτείνω την κυρία Ζουλί Λεσαντού, Ζουλή ως τέταρτη αντιπρόεδρο, υποψήφια. Y a t ε, Υπάρχει Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια για την εκλογή σας πρώτα απ' όλα. Θα ήθελα να προτείνω ο συντονιστής της ομάδας Renew Europe, τον κύριο Ζαν Jean-Christophe Ατχά, για τέταρτο αντιπρόεδρο. Μάλιστα, για τον τέταρτο αντιπρόεδρο έχουμε δύο υποψηφιότητες. Την κυρία Λεσοντού και τον κύριο από, την ομάδα Άλντε λέει η πρόεδρος. Ε, όχι και Άλντε. Α, ναι, ζητώ συγγνώμη, έχω μείνει λίγο πίσω. Ναι, εσείς ανανεώνετε. Το, το, μου είχε διαφύγει. Ε, συμφωνείτε, έχουμε δύο υποψηφίους. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε. Παρακαλώ. Πώς λέγεστε, Ολιβιέ λέγομαι. Από την ομάδα ID. Εγώ θα ήθελα να πω ότι αντίθετα με τους κανόνες ευγενίας αλλά και δημοκρατίας, Βλέπουμε εδώ ε, μια κοροϊδία, εμπεγμός. Ε, ε, ο εσωτερικός κανονισμός του Κοινοβουλίου τι ορίζει και δεν τον έχω γράψει εγώ. Οι μειονότητες θα πρέπει, οφείλουν να εκπροσωπούνται. Αυτό είναι υποχρέωση. Και με τη δεύτερη αυτή υποψηφιότητα η ομάδα μας, από ό,τι φαίνεται, θα στερηθεί εκπροσώπηση ε, στο Προεδρείο. Αυτό το θεωρούμε και το σκάνδαλο και παρακαλώ τους συναδέλφους να διορθώσουν αυτή την αδικία που θα δημιουργηθεί ψηφίζοντας την κυρία Λισαντού. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ολιβιέ. Νομίζω ότι ουδής ε, εδώ σε αυτή την Επιτροπή δεν δικαιούται να κάνει μαθήματα δημοκρατίας. Έχουμε δύο υποψηφίους Μπορεί ο καθένα να είναι υποψήφιο. Δύο υποψηφίου διαθέτουμε αυτή τη στιγμή. Εδώ στην Επιτροπή μα δέχεστε όλοι ε, να θέσουμε σε ψηφοφορία τα δύο ονόματα. Συμφωνείτε όλοι. Ωραία. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικώ. Η κυρία Λεσάντου και ο κύριο. Δέχεστε να είστε υποψηφία, μάλιστα. Ναι ή όχι. Ευχαριστώ όλες τις πολιτικές ομάδες. Ε, ομάδες, ε, όλες τις συνιστώσεις μάλλον της ομάδας μου ε, για την εμπιστοσύνη τους και με τιμή και ταπεινότητα δέχομαι αυτή την υποψηφιότητα. Κύριος Χόιτενς, έχετε το λόγο. Δέχεστε την υποψηφιότητα, αγαπητή Πρόεδρε, με πολύ μεγάλη τιμή. Θα υπηρετήσω εδώ ως αντιπρόεδρος, τέταρτος αντιπρόεδρος και δέχομαι την υποψηφιότητα. Έχουμε λοιπόν δύο υποψηφίους. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Έχετε όλοι τις κάρτες σας. Αν έχετε τις κάρτες σας όλοι. Άρχεται η ψηφοφορία. Να κάνουμε μια δοκιμαστική πρώτα. Ναι, ναι, μια στιγμή. Τεστ. Μια δοκιμαστική ψηφοφορία για να δούμε αν λειτουργούν τα μηχανήματα. Αν είστε όλοι χαρούμενοι, ε, να ψηφίσετε πράσινο, να πατήσετε το πράσινο το κουμπάκι. Και αν είστε δυσαρεστημένοι, το κόκκινο. Η δοκιμαστική ψηφοφορία είναι αυτή c'est le vert. Et Λοιπόν, ευχαριστημένη, πράσινο, δυσαρεστημένη, κόκκινο. Λήξεις ψηφοφορίας. Σαράντα. Είστε πανευτυχείς. Και οι δύο που δεν ξέρουν τι είναι σήμερα, λάει, ε, Λοιπόν, για το τέταρτο αντιπρόεδρο είναι απλή η διαδικασία. Το πράσινο θα είναι για την κυρία Λεσάντου. Το κόκκινο θα είναι για τον κύριο Χέιτενς. Εντάξει. Όποιος ψηφίζει πράσινο, ψηφίζει την κυρία Λεσαντέ. Όποιος ψηφίζει κόκκινο, τον κύριο Χέιτενς. Το καταλάβαμε όλοι. Αρχίζει λοιπόν η ψηφοφορία. Tout le monde a voté. Ψηφίσατε όλοι. Το ΕΛΚ έχει έναν υπεράριθμο. Ωραία αρχίσαμε. Α, όπως πάντα. Κάποιος ψήφισε ε, παραπάνω. Βγάλτε μια κάρτα. Allez, très bien. Τώρα είμαστε εντάξει. Λήξεις. 31 ε, ψήφισαν το, τον κύριο Χόιτενς, 16 την κυρία Λουσαντουέ. Κύριε Χόιτενς, ε, ε, ανακηρύσσετε τέταρτος αντιπρόεδρος. Έλατε κι εσείς στο Προεδρείο. Γι, Αγαπητοί συνάδελφοι, ραντεβού για την επόμενη συνεδρίασή μας στις 24 Ιουλίου στις 9 η ώρα το πρωί. Να έρθετε. Μετά οι συντονιστές, μόνο οι συντονιστές θα συνεδριάσουν την άλλη εβδομάδα στις 19 Ιουλίου. Αν δεν έχετε άλλες παρατηρήσεις αγαπητοί συνάδελφοι, κηρύσω το πέρα συνεδρίαση και σας ευχαριστώ.